και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για πέντε ε, ψηφίσματα, για πέντε προτάσεις ψηφίσματος για το Θιβέτ, ειδικότερα για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στις περιπτώσεις μοναχών. Λοιπόν, ψηφίζουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, είχατε όλοι την ευκαιρία να ψηφίσετε. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορίας το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο, εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, ψηφοφορία για έξι προτάσεις ψηφίσματος για τον Μπαχρέιν. Κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα συνολικά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με διαφορά. Και τέλος η υπόθεση της Ραφάνα Σέτ. Και πάλι ονομαστική ψηφοφορία, κοινή πρόταση ψηφίσματος. Ψηφίζουμε το συνολικά. Υπέρ. Μάλλον έναρξη και πέρας. Προφανώς εγκρίθηκε με σαφή πλειοψηφία. κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, ε, ε, θα έχουμε εξηγήσει ψήφων όσον αφορά την